ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ντάλι, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Την συζήτηση για την φαρμακοεπαγρύπνηση, κοινή συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Λίντα Μακάβαν, η μία έκθεση αφορά την τροποποίηση της οδηγίας και η άλλη την τροποποίηση του κανονισμού. Ξεκινώντας θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακάβαν για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η φαρμακοεπαγρύπνηση αφορά βέβαια την ασφάλεια των φαρμάκων και την παρακολούθηση της λειτουργίας του στην αγορά και την αντιμετώπιση δεχομένων παρενεργειών. Πριν από δύο χρόνια, εμεί ω Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνυπογράψαμε με την Επιτροπή μια μεγάλη μεταρρύθμιση και δεν περιμέναμε ότι δύο χρόνια αργότερα θα βρισκόμασταν να ξανασυζητούμε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό ήταν πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο Mediator στη Γαλλία που αποκάλυψε αδυναμίε όσα είχαμε ήδη αποφασίσει. Κύριε προτεραιότητα για μένα λοιπόν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, των τελευταίων αυτών εβδομάδων ήταν να ενισχύσω ιδιαίτερα το ρόλο του ρυθμιστικού φορέα στο σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης προκειμένου να ενισχύσω την ασφάλεια για τον ε, ασθενή. Ε, Ξετάζοντα ιδιαίτερα την υπόθεση με Mediator, προκύπτουν δύο ξεκάθαρα για μένα ζητήματα. Καταρχά, τα ζητήματα τη ασφάλεια είχαν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων αλλά δεν είχε παραπευθεί το θέμα για ε, εξέταση τυπική και είχε αφαιθεί η εταιρεία να διαχειριστεί μόνη της το θέμα με εμπορικά κίνητρα στις διάφορες χώρες. Δεύτερον, οι Ιταλικές αρχές είχαν ζητήσει μελέτη από τη Σερβιέ για την ασφάλεια του, φαρμάκου ήδη από το 2000. Γιατί υπήρχαν ακριβώς ανησυχίες περί παρενεργειών, αλλά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη. Δεν, είχε, ε, δεν ολοκληρώθηκε πριν να περάσουν 10 τουλάχιστον χρόνια και μάλιστα το μεταξύ λόγω της επαρή ε, κάποιου περιφερειακού υπεύθυνο φάρμακο στη Γαλλία είχε ήδη αποσυρθεί το φάρμακο. Έτσι λοιπόν με δεδομένο αυτό και τι παρατηρήσει μα από την υπόθεση Μερκατόρ, κάναμε, Μεντιατόρ κάναμε κάποιε σημαντικέ αλλαγέ. Δηλαδή χρειάζεται περισσότερη ε, ε, επιτήρηση μιας εταιρείας να αποφασίσει μόνη της αν αποσύρει ένα φάρμακο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι δυνατόν να της υποβάλλονται ερωτήσεις και να ελέγχονται οι όροι που τους οποίους αποσύρεται ένα φάρμακο. Δεύτερον, η αδίποτε ανησυχία περί της ασφάλειας των ασθενών θα αποτελεί σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό με έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα μπορεί μια χώρα να αποφασίζει μόνη της τι θα πράξει. Τρίτον, όταν απαιτείται μία ε, μελέτη ασφάλειας μετά τη χορήγηση της άδειας για το φάρμακο θα πρέπει αυτή να διεξάγεται. Ιδάλλως, φάρμακα τα οποία ε, είναι, για τα οποία εκκρεμεί μια μελέτη θα χαρακτηρίζονται με ένα μαύρο τρίγωνο και έτσι θα γνωρίζει το κοινό, ο ιατρικός κόσμος ε, ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και αυτό που ήταν εντυπωσιακό στην περίπτωση του Μεντιατόρ ήταν ότι δεν υπήρχε η σχετική εξουσία από πλευράς των γαλλικών αρχών να χαρακτηρίσουν δηλαδή, το φάρμακο ε, ως ύποπτο για επανεξέταση ενώ ήδη είχε χορηγηθεί η σχετική άδεια για τη διάθεση του εμπόριο. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να επισημάνω ακόμη ζητήματα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, κύριε Επίτροπε, και με το λεγόμενο black box, δηλαδή την ε, τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με αυτές που προκύπτουν στο φυλάδιο για τον ασθενή. Είχατε πει κύριε Επίτροπε ότι στα δύο αυτά ζητήματα θα μου απαντήσετε και ελπίζω ότι θα απαντήσετε λεπτομερώς. Και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους ε, τους σκιώδεις ηγητές που είναι εδώ παρόντες για όλη τη σκληρή δουλειά που κάνανε τις προσπάθειές τους και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Προεδρία της Δανίας την Επιτροπή, την Προεδρία του Συμβουλίου, γιατί η Προεδρία του, Συμβουλίου ήταν εκείνη η οποία βοήθησε να προχωρήσει η δουλειά αυτή ταχύτατα, ώστε με τη συμφωνία να έχουμε προχωρήσει πριν από το καλοκαίρι, ώστε ε, να προχωρήσει σε υλοποίηση συμφωνία αυτή μαζί με τις λοιπές αλλαγές στην, ε, διάταξη, στην νομοθεσία για τη ε, φαρμακοεπαγνήμιση. Ευχαριστώ κύριος Δαλή. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να ξεκινήσει η πρώτη ανάγνωση της συμφωνίας για τα θέματα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία την κυρία Μακάβεν φυσικά η οποία διευκόλυνε κατά πολύ θα έλεγα να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση γρήγορα. Το λεγόμενο stress test, το έλεγχος ακραίων καταστάσεων και συνεπειών, περιλαμβάνεται στην πρόταση. Η σημερινή πρόταση ενισχύει την διαφάνεια και τις υποχρεώσεις αναφοράς. Υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων που θα υποστούν περισσότερους ελέγχους έτσι ώστε να αποδειχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης τους. Απαιτείται επίσης ε, και ε, προβλέπεται να υπάρξουν περισσότερες εξηγήσεις για την απόσυρση ενός προϊόντος από την ε, εταιρεία τη φαρμακευτική. Πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι, ιδιαίτερα όταν τίθενται θέματα ασφαλείας. Η εμπιστοσύνη των ασθενών στα φαρμακευτικά προγράμματα είναι κάτι το απαραίτητο και μπορούμε να την πετύχουμε και να την διατηρήσουμε εφόσον οι ασθενείς σέβονται και εμπιστεύονται το σύστημά μας. Η πρόταση την οποία θα υιοθετήσει αύριο το Κοινοβούλιο ελπίζω θα ενισχύσει τις νομικές ρυθμίσεις γύρω από το θέμα της επαγρύπνησης στα φάρμακα και ελπίζω πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δηλώνει ότι στον Ιούνιο του 12 ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για την εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων για την φαρμακοεπαγρύπνηση ε, και για τις πιθανές αλλαγές των νομικών ρυθμίσεων που είχαν αποφασιστεί το 2010 τελείωσε η διαδικασία ή τελειώνει στις 15 Σεπτεμβρίου και ε, θα εξετάσουμε την νομική κατάσταση του θέματος πριν κάνουμε νέες προτάσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να θεωρούμε το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης σαν προτεραιότητα και θα καταθέσουμε την νομική μας πρόταση στο Κοινοβούλιο ε, και στο Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ τον κύριο Ντάλι. κυρία Γιούζο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι έκανε πολύ μεγάλη δουλειά η κυρία εισηγήτρια Μακάβαν, καθώς επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές, για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Πράγμα πολύ σημαντικό για την έναρξη σε ισχύ του, του κανονισμού ε, σε σχέση με το 2010 αυτό ο κανονισμός έπρεπε να αναθεωρηθεί και θα έπρεπε λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα πρόσφατα αυτά γεγονότα που τα γνωρίζουμε όλοι που έδειχναν ότι υπάρχει ένα κενό και έπρεπε να επανορθωθεί η κατάσταση για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό με συγκεκριμένα σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν σε σχέση με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Γι' αυτό εφ' εξής, όπως αναφέρθηκε θα έχουμε σε σχέση με την ε, εμπορία ενός ε, φαρμάκου που δεν θα ε, έχει την παράταση θα έχει την υποχρέωση να μπορέσει να αποσαφηνίσει τους λόγους που οδηγούν στην λήξη της εμπορίας αυτού του προϊόντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό προς όφελος των καταναλωτών ώστε να μπορέσουν να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί λόγοι για αυτή την κατάσταση πραγματικότητα και επιπλέον σε σχέση και με τα όσα συμβαίνουν σε μια τρίτη χώρα θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση η διαφάνεια και η ασφάλεια θα πρέπει να διασφαλιστούν λαμβάνοντας υπόψη και την, ε, το, διαφανή, το διαφανές πλαίσιο για τα φάρμακα. Δεύτερη πτυχή που είναι σημαντική είναι ότι όλα τα ε, φάρμακα τα οποία θα ε, τίθενται στην αγορά αμέσως θα εντάσσονται σε ένα κατάλογο προϊόντων που θα πρέπει να υφίστανται αυτή τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Επίσης ε, η φαρμακοεπαγρύπνηση έχει θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει και γι' αυτό πρέπει η Ολομέλεια, οι Ευρωβουλευτές να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Κυρία Κάρενμπαχ, και εγώ από πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Λίντα Μακάβαν και τους σκιώδεις εισηγητέ και εισηγήτριε. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έδρασε ταχύτατα σε σχέση με το 2010 για κάτι το οποίο θεωρούσαμε αποτελεσματικό που όμως ε, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματικό και μπορέσαμε να διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα και το κενό, το χάσμα αυτό έπρεπε να καλυφθεί. Χρειαζόμαστε τη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε τον γοργό τρόπο δράση, ε, την ταχύτητα. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα φάρμακα. Χρειαζόμαστε επίση και την εμπιστοσύνη στο συνολικό σύστημα από πλευρά των πολιτών. Πρέπει η ίδια η συνεργασία να διασφαλιστεί για τα φάρμακα τα οποία ε, κυκλοφορούν στην Ευρώπη, ώστε υστερότερα να μπορούμε να επαγρυπνήσουμε, να υποπτεύσουμε αν υπάρχουν παρενέργειες ή αν υπάρχουν βλαπτικές ε, παρενέργειες και έτσι στη συνολική ευρωπαϊκή αγορά άμεσα να υπάρχει ταχύτατα ενημέρωση για τέτοια συμβάντα. Ένα ε, φάρμακο να μην μπορεί απλά ε, και παραβίστο να αποσύρεται από την αγορά αλλά να αποκαλύπτονται οι λόγοι για τους οποίους αποσύρεται από την αγορά. Χρειάζεται ταχύτατα η διαφάνεια και η φαρμακοεπαγρύπνηση. Χρειαζόμαστε στενή συνεργασία με τους ασθενείς αλλά επίσης και με το προσωπικό στον τομέα των υγειονομικό. Πρέπει επίσης ε, να πούμε ότι μόνο τότε μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί αν όλοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συγκλίνουν και να διαχέονται με το σωστό τρόπο. Μόνο τότε μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν μπορούν οι ασθενείς να κατανοήσουν με εύληπτο τρόπο περί πρόκειται. Και όπως ανέφερε και η κυρία Λίντα Μακάβεν από πλευρά των χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων που θα δημιουργηθούν να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ την κυρία Μακάβαν για την προσπάθειά της και την καθοδήγησή της και να ευχαριστήσω και τις πολιτικές ομάδες που μας επέτρεψαν να συμφωνήσουμε δύο χρόνια μετά την υπόθεση Μεντιατόρ στη Γαλλία που αποκάλυψε όλα τα κενά που υπήρχαν στα πλαίσια της φαρμακοεπαγρύπνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αποδεικνύουν σήμερα ότι όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών μπορεί να αναλυθεί ταχύτατα η δράση που απαιτείται για την αντιμετώπιση της. Προετοιμάζεται λοιπόν η μεταρρύθμιση του πλαισίου που υιοθετήθηκε το 2010 έτσι ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά ή που αποσύρονται από την αγορά. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η υποχρέωση για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τους λόγους για την απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά και δεύτερον η θέση σε λειτουργία της αυτόματης διαδικασίας έρευνας όταν δημιουργούνται υποψίες. Έτσι θα διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος φαρμακοεπακρύπνησης, θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και την κατανόηση της κατάστασης από πλευράς των πολιτών. Έχουμε ευθύνε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνε αυτές για να προσαρμόσουμε το σύστημά μας και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητά του. Απαιτείται να υπάρξουν και οι απαιτούμενοι πόροι οι οποίοι θα διασφαλίσουν στην υπηρεσία την Ευρωπαϊκή για τα φάρμακα τη νέα αποστολή της με εύρυθμο τρόπο. Θα γίνει νομίζω και πρέπει η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν. Η κυρία Γιανακουδάκη έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ασφάλεια των ασθενών πρέπει πάντοτε να είναι η κυρία μας προτεραιότητα. Πρόσφατες ε, πληροφορίε πληροφορίες σε σχέση με το φάρμακο Μεντιατόρ οδήγησε σε θάνατο πολλού ε, ασθενεί και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνονται οι ασθενεί για τις παρενέργειες του φαρμάκου, κάθε παρενέργεια. Πρέπει λοιπόν να κλείνουν τα παραθυράκια και πρέπει να είναι υποχρεωμένε οι ε, φαρμακο, φαρμακευτικές επιχειρήσεις να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ένα φάρμακο στην δημοσιότητα. Με ικανοποίηση βλέπω ότι η έκθεση έτυχε ταχείας και αποτελεσματικής επεξεργασίας. Χρειάζεται ε, βεβαίως αλλαγή στην νομοθεσία. Ε, η ασφάλεια των ασθενών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και έστω και αν χρειαστούν περαιτέρω τροποποίηση, είναι απαραίτητο τώρα να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα για να θεθεί σε εφαρμογή αμέσω. Και συγχαίρω την κυρία Μακάβων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ρώση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Λίντα για την προσπάθεια που έκανε. Με την θέση σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων θα ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των φαρμάκων. Οι στόχοι στρατηγική της νέας οδηγίας και του νέου κανονισμού συμβαδίζουν με τις ρυθμίσεις ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον φαρμακευτικό τομέα. Πρέπει να ελέγχεται καλύτερα η υγεία των πολιτών, να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Είναι απαραίτητο για την προστασία των πολιτών να ενισχυθούν τα συστήματα της φαρμακοεπαγρύπνησης, μια καλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης του συστήματος έτσι ώστε να κριθεί η ανεκτικότητα ενός φαρμάκου σε σωστό και ρεαλιστικό ε, πλαίσιο χρήσης. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Ο κύριος Μαστάλκα, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους εκείνους τους συναδέλφους που υποστήριξαν και ευχαρίσαν την κυρία Μακάβαν για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε το μεγάλο έργο σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Με ικανοποίηση και χαρά βλέπω ότι είχαμε τριμερή διάλογο ικανοποιητικό που μπόρεσε σε πρώτη ανάγνωση να φέρει αποτελέσματα και είμαι πεπισμένο ότι οι τροποποιήσεις ε, στην νομοθεσία αυτή θα επιφέρουν καλύτερη προστασία για τον ασθενή στην Ευρώπη. Χρειάζεται και εξασφαλίστηκε καλύτερο τονισμό μεταξύ των κρατών μελών και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε τέτοιου είδους σκάνδαλα όπως αυτό του Μεντιάτορ στο μέλλον να τα αποτρέψουμε, να τα αποφύγουμε. Η νομοθεσία αυτή ε, δεν μπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν υλοποιηθεί σωστά, εάν δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει. Η οικονομική κρίση ξέρουμε ότι ε, συνεπιφέρει πολλές περικοπές και γι' αυτό απαιτείται να μεριμνήσουμε ώστε τα κατάλληλα όργανα, οι φορείς ε, στα κράτη-μέλη αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη οικονομική πρικοδότηση αλλά και το προσωπικό πάνω απ' όλα το οποίο θα επιτελεί το έργο αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Μαστάλκα και τώρα ο κύριος Σόπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ η φαρμακοεπαγρύπνηση και ιδιαίτερα η παρακολούθηση της λειτουργίας των φαρμάκων μετά την αδειοδότηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία της υγείας του ασθενούς. Πολλές φορές κάποια στοιχεία προκύπτουν για ένα φάρμακο μετά τη διάθεσή του στην αγορά και έτσι χρειάζεται επιπλέον η πρόσθετη επαγρύπνηση, παρακολούθηση του φαρμάκου και μελέτες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται με ένα μαύρο συμβολό πάνω στο κουτί το φάρμακο που βρίσκεται σε αυτή τη φάση της επανεξέτασης. Και πρέπει επίσης να ε, καθίσετε γνωστό το για ποιο λόγο όταν αποφασίσει μια, επι... μια φαρμακευτική επιχείρηση να αποσύρει ένα φάρμακο από την αγορά να ενημερώνει τους λόγους για τους οποίους το πράττει αυτό. Δεν μπορεί να μην ενημερώνεται ο φαρμακοποιός ή ο ιατρός για τους λόγους για τους οποίους αποσύρεται ένα, ένα φάρμακο και αυτό γιατί πρέπει να γνωρίζουν ε, ακριβώς ποιοι είναι οι λόγοι. Ευχαριστώ κύριος Λύση, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που συνέβησαν στο σκάνδαλο. Στην περίπτωση με τώρα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι, πόσα είναι τα θύματα, από 500 έως 2.000 αναφέρεται, αλλά όπως και να είναι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη. Ε, λέγεται ότι έπραξε κακώς η επιχείρηση η ίδια, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και προβλήματα ως προς την νομοθεσία, κενά δηλαδή νομοθετικά. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερως που η κυρία Μακέβαν, η Λίντα, αλλά και η σκιώδη συγγήτρια κυρία Αγιούσο και ο επίτροπος κύριος Δάλη ε, επεξεργάστηκαν όπως επεξεργάστηκαν την πρόταση και την προώθησαν μέχρι την αναθεώρηση αυτή. Είναι σημαντικό στο μέλλον να εξηγείται γιατί αποσύρεται από την αγορά ένα φάρμακο όταν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια και είναι απαραίτητο να ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους επακριβείς πληροφορίες ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Η κυρία Κέμπερ και ο υποφαινόμενος επιπλέον των όσων είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτουμε μια τροπολογία για το λεγόμενο κοιτίο δεδομένων για τα φάρμακα. Και θα έλεγα ότι πρέπει να ονομάζεται στα αγγλικά όχι black box, μαύρο κουτί, αλλά ε, drug fact box, δηλαδή κοιτή δεδομένων για τα φάρμακα. Είναι μια πρόταση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίμησε, αν και εγώ νομίζω ότι δεν ε, δίνει τον κατάλληλο συμβολισμό και έννοια η λέξη, η φράση μαύρο κουτί. Εν πάση περιπτώσει όμως θα ήθελα να αναφερθώ στο σύστημα των ΗΠΑ με αυτό το κοιτίο δεδομένων που ισχύει στις ΗΠΑ, αποδεδειγμένα με καλά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι είναι πολλές φορές περίπλοκα τα στοιχεία που καταγράφονται στα δελτία των φαρμάκων ε, στο φυλάδιο που συνοδεύει το φάρμακο ε, και θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ειδών, δύο κατηγορίες ε, ασθενών. η μία κατηγορία δεν διαβάζει καν το φυλάδιο αυτό, το πετάει απλώς στα σκουπίδια. Ενώ η το διαβάζει πολύ προσεκτικά και τρομοκρατείται από όλες τις πιθανές παρενέργειες και επιπλέον ανεπιθύμητες ε, ε, συνέπειες, επενέργειες που μπορεί να έχει το φάρμακο. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, υπογραμμίζονται οι σημαντικές πτυχές βεβαίως. Επίσης όμως θα πρέπει και στο φυλάδιο να υπογραμμίζεται ιδιαίτερως ότι θα πρέπει να καταναλώνετε, να προσλαμβάνετε το φάρμακο όπως ακριβώς το έχει χορηγήσει ο γιατρός με βάση τη συνταγή. Ιδιαίτερα για τα αντιβιωτικά είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε με μεγάλη ακρίβεια συνταγή. Αυτή λοιπόν η μέθοδος με το, με το κοιτίο δεδομένων ε, στις ΗΠΑ έχει φέρει καρπού, έχει υποδεδειγμένα λειτουργήσει καλά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το κύτταρο δυνατό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια ακριβή πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπένοβα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Stress tests ιδιαίτερα στον τομέα της φαρμακοεπαγνύπνησης είναι σημαντική υπόθεση. Διαπιστώθηκε ότι στο νομικό σύστημα της ΕΕ υπάρχουν μεγάλα κενά και πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να υφίστανται τέτοιου είδους κενά. Για το Μεντιάτορ το φάρμακο αυτό, το φάρμακο είχε άδεια κυκλοφορία σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες πληροφορίες έδειχναν ότι υπήρχαν παρενέργειας ε, σε σχέση με αυτό το φάρμακο ήδη χρόνια πριν. Παρόλα αυτά συνταξιο... συνταγογραφούσαν οι γιατροί αυτό το φάρμακο και συνέχιζαν να το παράσχουν στους ασθενείς. Εκατομμύρια άτομα το χρησιμοποίησαν. Υπολογίζεται ότι μέχρι 2.000 άνθρωποι αποβίωσαν λόγω της ε, λήψης της χρήσης αυτού του φαρμάκου διάφορες αρχές και διάφορες συναντήσεις ε, ειδικών οδήγησαν σε συζητήσεις για αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά όμως δεν ελήφθη καμία σχετική απόφαση για αυτό το φάρμακο. Αυτό τι σημαίνει. Σε επίπεδο ΕΕ δεν έγινε έλεγχος ε, αυτού του φαρμάκου. Δεν αντέδρασαν οι ρυθμιστικές αρχές. Όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν ότι τα φάρμακα σε σχέση με την εμπορία τους πρέπει προηγούμενα να ελέγχονται σε ε, ιδιαίτερα προσεκτικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και πρέπει προ όφελο τη υγεία των πολιτών αυτέ οι αλλαγέ να διασφαλιστούν το δυνατόν ταχύτερα. Και θέλω να ευχαριστήσω του κοιόδης εισηγητέ για τη συνεργασία του. Η κυρία Ρή, ευχαριστώ. Oh, ευχαριστώ. Ποτέ δεν θα γνωρίσουμε τον αριθμό των νεκρών από το φάρμακο Mediator αλλά στην ουσία το έδιναν περισσότερο για να κόβει την όρεξη. Δυστυχώς υπήρξαν πάρα πολλά θύματα. Χρειάστηκε να περιμένουμε το 2009 για να αφαιρεθεί η κυκλοφορία του φαρμάκου, να απαγορευτεί το φάρμακο από την κυκλοφορία, ενώ είχε κοπεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ισπανία και την Ιταλία. Είναι απαραίτητες οι αλλαγές αυτές λοιπόν λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν ένα προϊόντα τα οποία χορηγούνται εκτός του συστήματος των συνταγών. Ε, οι αδυναμίες του συστήματος που ψηφίστηκε, που αποφασίστηκε και πριν δύο χρόνια είναι σαφής πλέον ε, πρέπει να ορίζονται οι λόγοι για τους οποίους μια εταιρεία φαρμακευτική αποσύρει ένα φάρμακο από την αγορά ή δεν ανανεώνει την άδεια κυκλοφορίας του πρέπει να ξεκινάει η κατεπίγουσα διαδικασία όταν οι ιατροί θεωρούν ότι η λήψη του συγκεκριμένου φαρμάκου δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των ασθενών τους για να λειτουργήσει όμως σωστά το σύστημα αυτό της επαγρύπνησης πρέπει οι ευρωπαϊκές αρχές και η υπηρεσία του Λονδίνου να λειτουργήσουν σωστά και να είναι ανεξάρτητες από τους εμπορικούς εταίρους του τομέα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές γιατί πράγματι οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΜΕΗ Υπηρεσία για τα Φάρμακα θα αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την ασφαλή κυκλοφορία των φαρμάκων. Το θέμα είναι η εμπορική άδεια κυκλοφορίας η οποία θα χορηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης υποχρέωση σωστής ενημέρωσης. Η γαλλική περίπτωση δείχνει ότι για πάρα πολλά χρόνια οι ευρωπαϊκές αρχές δεν ήταν σε θέση να απαγορεύσουν το φάρμακο αν και κάποια μεμονωμένα κράτη-μέλη είχαν αποσύρει ουσιαστικά την κυκλοφορία ε, του φαρμάκου. Ε, συνειδητοποιούμε το ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν τεράστια εξουσία, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ματίας, μισή λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω την φωνή μου σε εκείνα τα σχόλια των συναδέφων που συνεχάρισαν την εισηγήτρια Λίντα Μακάβεν για την εξαιρετική δουλειά που έκανα οι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη νέα ρύθμιση θα είναι πολύ πιο ασφαλείς σε σχέση με τον κανονισμό και ιδιαίτερα σε σχέση και με τις προτεραιότητες που δίνουμε. Με όλα αυτά σε σχέση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα που παρατήρησα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Το πρώτο αφορά την οικονομική κρίση που βλέπουμε ότι πλήττει τις ε, υγειονομικές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, δρατώμενοι της ευκαιρίας, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε η οικονομική κρίση να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην φαρμακοεπαγρύπνηση σε σχέση με την ενημέρωση και πληροφόρηση των ε, ασθενών και να καθυστερήσουμε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα η κρίση. Με κάθε μέλημα και προσοχή σε σχέση με τα νέα φάρμακα δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να δεχθούμε να υπάρχουν υπάρχουν κενά και προβλήματα. Αυτό είναι αναγκαίο διότι από το 2010 βλέπουμε ότι είχαμε κάποια ζητήματα με αυτή την οδηγία και φτάσαμε στο 2012 για να μπορέσει να γίνει κάτι. Το 2010 και σήμερα το 2012 πρέπει να πούμε ότι αυτό πια αρκεί και στην ε, ε, Ελλάδα και σε άλλες ε, χώρες υπάρχουν προβλήματα με τα φάρμακα και την, τα όσα δίνονται στους ασθενείς. Πρέπει εδώ το πειραματικό αυτό εργαστήριο, το φαρμακευτικό εργαστήριο να λάβει υπόψη αυτά τα προβλήματα και είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για την υγεία των κατοίκων μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρόσετ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Euh, Ευχαριστώ. Επίτροπε, συγχαίροντας τον στην εισηγήτρια, θα ήθελα να συγχαρώ και τον Επίτροπο Ντάλι για την ανταπόκρισή του στην περίπτωση του Μεντιατόρ. Λόγω ακριβώς αυτής της ανταπόκρισης έγιναν τα διάφορα τεστ και τα οποία προτείνονται και στα πλαίσια ακριβώς των προτάσεων για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Αυτά τα τεστ ακραίων καταστάσεων και αντιδράσεων έδειξαν ότι υπάρχουν αδυναμίες στην ομοθετική μας ρύθμιση και σήμερα όταν προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στις αδυναμίες που έχουμε παρατηρήσει το κάνουμε ενισχύοντας τη διαφάνεια, ενισχύοντας την επικοινωνία για την ασφάλεια των τροφίμων. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ένα θέμα θα έλεγα αδυναμίας. Λυπάμαι γιατί η νέα αυτή νομοθεσία δεν ασχολείται με το θέμα της ειδική κατηγορίας συνταγών, συνταγολόγησης, ειδική συνταγολόγησης η οποία αντιπροσωπεύει μέχρι το 15% του συνόλου της συνταγογράφησης αυτού του είδους λοιπόν οι συνταγογραφήσεις μπορεί να είναι χρήσιμες αλλά παρουσιάζουν και κάποιο είδους ε, κινδύνους ε, γιατί μπορεί να γίνονται εκτός έγκρισης των αρχών στον τομέα της υγιεινής. Πολλές φορές ε, δεν θα υπάρχει καταγραφή των συνεπειών της χρήσης αυτών των ουσιών από πλευρά των ειδικών, κάτι το οποίο δεν θα επιτρέψει στους τομείς αυτούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το να ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να οδηγηθεί στο συγκεκριμένο τομέα με τη, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για αυτού του είδους της ειδικού τύπου συνταγογραφήσεις είναι κάτι που έπρεπε να ζητηθεί λοιπόν και έτσι να καλύψουμε κάποιες ειδικές θεραπευτικές ανάγκες. Εν πάση περιπτώσει η περίπτωση του φαρμάκου Μεντιατόρ χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και διέφυγε ελέγχου η χρήση του. Αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον. Κυρία Βάισμπεργκερ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Μακέιβαν για την πολύ καλή της δουλειά, την πολύ καλή έκθεση. Μια ουσιαστική φαρμακοεπαγρύπνηση και προστασία του πολίτη ταυτόχρονα σημαίνει καλύτερη ασφάλεια για τον ε, ασθενή. Βλέπουμε με την υπόθεση Μεντιάτορ ότι κατέστη απαραίτητο πολύ γρήγορα να κλείσουν κενά στην νομοθεσία. Υπήρχαν δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες μπορούσαν να αποσύρουν για δικούς τους λόγους ένα φάρμακο από την αγορά. Ε, με το νέο σύστημα λοιπόν ενημερώνονται τα κράτη-μέλη και σε τελευταία ανάλυση αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προσοχή του πολίτη και του ασθενούς. Απαραίτητο είναι να είναι πιο ευανάγνωστα πιο ξεκάθαρα τα κείμενα στο φυλάδιο που συνοδεύει το φάρμακο γιατί για πολλούς ασθενείς είναι ε, πολύ δυσ... Ε, ε, δυσνόητο, είναι αδιαφανές, ασαφές, δεν καταλαβαίνει δηλαδή ο ασθενής τη διαβάζει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ε, οι απαραίτητες πληροφορίες ε, για τις ε, παρενέργειες, όχι όμως σε βαθμό που να τρομάζουν τον ασθενή και να μην τολμάει αυτός να το πάρει. Άρα όπως είπε και ο κύριος Λίσε, πρέπει να είναι πιο σαφές το κείμενο, πρέπει να υπάρχει και ένα κοιτίο δεδομένων για το φάρμακο σε μια απλή κατανοητή γλώσσα και ε, να δίνονται πρακτικές πληροφορίες και οδηγίες για το φάρμακο. Θα ήθελα επίση ε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι και η Επιτροπή με τον κύριο Νταλή μα πρόσχεται ότι θα μεριμνήσει για την ε, πιο σαφή διατύπωση και κατανοητή διατύπωση των οδηγιών και του φυλαδίου του φαρμάκου. Δεν ξέρω αν εδώ, εφόσον εδώ ο κύριος Νταλή, αν είναι σε θέση να μας πει ότι έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδέες και να μας τις εξηγήσει ή όχι. Πάντως θεωρώ ότι έχουμε πραγματοποιήσει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ασφάλεια του ασθενούς, αν καταφέρουμε να διατυπώσουμε ένα φυλάδιο του φαρμάκου πιο σαφές, πιο ευανάγνωστο, πιο κατανοητό. Ευχαριστώ κύριο Μπάνκι για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λίντα Μακάβεν για την ταχεία, ταχύτατη εργασία της με αποτελεσματικό τρόπο στη σύνταξη της εκθεσής της. Πρόκειται για ένα πεδίο τεράστιας σημασίας που αποδεικνύει ότι σε αυτό το θέμα είμαστε ικανοί ως Ευρωκοινοβούλιο να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευελπιστώ ότι αυτή η συνεργασία θα δώσει τον καρπό της και θα καρποφορήσει θετικά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο ε, πρέπει να τύχει της προσοχής μας. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στην ε, ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους για την ασφάλεια φαρμάκων υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και οι χειρότερες ε, καταστάσεις είναι εκείνες που δείχνουν ότι όπως είπε ο κύριος Λίσε και άλλοι ότι είναι και προβλήματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα. Οι περισσότεροι ασθενείς ούτε διαβάζουν καν τις οδηγίες για τη χρήση ενός φαρμάκου. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ασθενών στα φάρμακα, αντιδρώντας άμεσα και αποτελεσματικά σε τέτοιες ελλείψεις και τέτοια προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένα φάρμακα. Όταν πριν από κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, είχαμε τα προβλήματα του ΙΤΑ ε, ε, 1 νι ε, του βακτηριδίου αυτού και της γρήπης που προκαλούσε είχαμε και προβλήματα στην Πολωνία και είχαν αναφερθεί στην Πολωνία τα επιχειρήματα να μην χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια ότι δεν ήταν ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια και διότι δεν είχαν αξιολογήσει και σωστά τους κινδύνους. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο προηγούμενο παράδειγμα. Αντιδρώντας άμεσα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών μας πρέπει να αφήνουμε κατά μέρο τις πολιτικές διαφορές και να συνεργαζόμαστε ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτή η έκθεση αποτελεί απόδειξη αυτής της αρχής. Όταν όλοι συνεργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία κυρία Τούρνεν-Χόεσταϊν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θέλει να αναθεωρήσει την οδηγία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τα φάρμακα που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν φυσικά πολύ μεγάλη σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ε, για τον πολίτη ότι τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει στο ίντερνετ ή στο φαρμακείο θα είναι και ασφαλή. Και ναι, τώρα αναθεωρείται η οδηγία και ο κανονισμός για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρόκειται για ένα βήμα ορθό προς τη σωστή κατεύθυνση αναμφιβόλα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και καλύτερη επικτήρηση και για τα άλλα προϊόντα στις αγορές, γιατί πολλές είναι οι επικίνδυνες ουσίες που κυκλοφορούν στις αγορές μας, ε, χωρίς να χορηγούνται ε, οι πληροφορίες στον πολίτη που θα του εξηγήσουν ε, ποιο φάρμακο μπορεί να είναι επικίνδυνο, τι θα πρέπει να αποφεύγει, από πού δεν θα πρέπει να αγοράζει. Μιλάμε για κίνδυνο για την ε, δημόσια υγεία, για την υγεία του ανθρώπου, για τη ζωή ακόμα των ε, συμπολιτών μας, ενώ πολλές φορές δεν γνωρίζει ο πολίτης ε, τα στοιχεία, τα δεδομένα όταν λαμβάνει ένα φάρμακο, τι συνέπειες μπορεί να έχει. Και πολύ σωστά επισημαίνει ο κύριος Λύση ότι χρειάζεται μια ευανάγνωστη ενημέρωση, ένα κοιτίο δεδομένων μια πρωτοβουλία πολύ καλή, η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση για τον καταναλωτή, εφόσον καταστεί υποχρεωτική η ορθή ενημέρωση για τις ενέργειες παρενέργειες ε, μιας ουσίας. Τώρα θα ήθελα κύριε Επίτροπε να ρωτήσω σε πόσες γλώσσες δεξάγεται η ε, διαβούλευση αυτή στην οποία αναφερθήκατε και απευθύνεστε και σε πολίτες που ενδεχομένω δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Ε, Πρόεδρε, κύριε Μικολάσιτ, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί όλοι συμφωνούμε πιστεύω εδώ ότι οι πληροφορίες για το καταναλωτή ε, σχετικά με τα φάρμακα πρέπει να βελτιωθούν, να καταστούν πιο ευανάγνωστες και βέβαια αυτό εσύ και για τα φάρμακα για τον καταναλωτή, για τις οδηγίες χρήσεως μέσα στο, στη συσκευασία που πρέπει να είναι επανάγνωστες και ορθές. Ωστόσο ερχόμαστε και στο ουσιαστικό ερώτημα κυρία Μακέβαν και θα ήθελα να τη συγχαρώ τη συνάδελφο διότι ε, πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα πρόοδου εξασφαλίζοντας ε, την ε, αναθεώρηση της νομοθεσίας αυτής έτσι ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τον ασθενή. Γιατί πολλές είναι περιπτώσεις όπου δίδεται ε, σε έναν ασθενή ένα φάρμακο προκειμένου να θεραπευτεί αυτός από μια νόσο, αλλά το φάρμακο το ίδιο του προξενεί πολλά προβλήματα με παρενέργειες έως και θάνατο. Αυτό το είδαμε στην περίπτωση του Mediator σε φάρμακα που, αφορούσαν τον διαβήτη συγκεκριμένα ή την καταπολέμηση της ε, ανορεξίας επίσης και αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία και την επιτυχία στο έργο σας. Κύριε Πασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε τις ρυθμίσεις του τομέα της επαγρύπνησης στη χρήση των φαρμάκων. Έτσι θα μειώσουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν. Είναι απαραίτητο επίσης οι οδηγίες χρήσης να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι κατανοητές. Και έτσι και οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση με πιο απλό και γρήγορο τρόπο. Δρώντας με τον τρόπο αυτό περιπτώσεις όπως η της του Μεντιατόρ δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Είναι βασικό να υπάρχει διαφάνεια στον τομέα της χρήσης των φαρμάκων για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρόιτεβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όλοι χαιρετίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε στην τραγική αυτή περίπτωση του φαρμάκου Mediator και ότι υπήρξε η υποχρέωση σε σχέση με την απόσυρση αυτού του φαρμάκου από την αγορά και ο συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων ενισχύθηκε. Όμως θα πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη για την τους λόγους, την αποκάλυψη των λόγων ε, για τους οποίους αποσύρεται ένα φάρμακο από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν διαπιστώνται προβλήματα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αμέσως θα πρέπει να προχωρούμε στη λήψη αναγκαίων μέτρων και στην ε, αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε παρό, να μην υπάρχουν κενά και παρόλη την νομοθεσία να μην γίνεται τίποτα όπως συνέβη στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταλή έχει τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, και κύριοι. Με ιδιαίτερα ευγνώμονε προ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη στην ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για τη μεταρρύθμιση στην φαρμακοεπαγρύπνηση. Όσον αφορά το μαύρο κουτί που αναφέρει η κυρία Μακέβαν, γίνεται αυτή τη μελέτη για την αξιολόγηση τη προσθέμενη αξία και των πληροφοριών που μπορεί να προσφέρονται στο λεγόμενο κοιτίο ε, στοιχείων για το φάρμακο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκου, με τις αρμόδιες εθνικές αρχές αλλά και με οργανώσεις και φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εκπροσωπούν καταναλωτές, ασθενείς, γιατρούς, φαρμακοποιούς, ασφαλιστές και την βιομηχανία του φαρμάκου. Γίνεται αυτή η μελέτη λοιπόν και η έκθεση για, την, για το ευανάγνωστον που ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους μήνες, ε, μέχρι τα μέσα του 2013 η σχετική έκθεση. Δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε, όπως υπόθηκε στην ε, οικονομική κρίση, να διατρίξει, να διαρρήξει το σύστημα προστασίας του ασθενούς και του καταναλωτή, ιδιαίτερα στα φάρμακα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς ένα από το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία. Έτσι λοιπόν, προσβλέπουμε στην υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας, στην υλοποίησή της, στην εφαρμογή της και στην εξασφάλιση για τον ασθενή και τον πολίτη ως το δυνατόν πιο σαφούς νομοθεσίας, ξεκάθαρης νομοθεσίας και παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακέιβαν, έχετε εσείς τον τελευταίο λόγο. Κύριε Μακέβαν, θέλω απλώς να απαντήσω στην κυρία Γκροστέτ ότι συμφωνώ πως η χρήση των ε, φαρμάκων πέραν της προβλεπόμενης ε, χρήσεως είναι πολύ σημαντικό ε, στοιχείο και πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερος. Για το κοιτίο δεδομένων έχει δίκαιο ο κύριος Λύς, είναι πολύ λεπτομερείς η ε, κατάλογη των ε, χαρακτηριστικών των φαρμάκων μέσα στο δελτίο αυτό, στο φυλάδιο το οποίο χορηγείται στο κοιτίο. Είναι σχεδόν σαν να διαβάζει κανείς ε, μια σύμβαση που έχει συντάξει δικηγόρος με πολλές υποσημειώσεις και υποπαραγράφους και είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβει κανείς. Θα ήθελα ιδιαίτερος όμως εγώ να ευχαριστήσω το προσωπικό του γραφείου μου που με έχει βοηθήσει ιδιαίτερος και ιδιαίτερα την βοηθό μου που δυόμιση χρόνια τώρα ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα ήθελα δηλαδή να αποτίσω φόρο τιμή σε όλους εκείνους, τη μου τη βοηθό αλλά και σε όλους τους βοηθούς μας και συνεργάτες μας που έχουν ε, τόσα πολλά προσφέρει στην προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακέβαν. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι και έτσι ε, αύριο αρχίζει 8.30 η συζήτηση μέχρι